Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζω τους αγαπητούς μας φιλοξενούμενους, Άφετ και τους συναδέλφους αντιπροσωπείας, Είχαμε έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας ΑΦΕΤ για τα Δυτικά Βαλκάνια. Καλωσορίζουμε και τους φιλοξενούμενους μας, τον κύριο Γκράμο Ρούτσι, Ντάνις Βίτζιτς, Γκλάουκ Κονιούφτσα, Ιβαν Τάλατ Τζαφέρι και την κυρία Κόικοβιτ, που ηγούνται των κοινοβουλίων των διαφόρων χωρών. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους που είναι παρόντες, για τους οποίους το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων τους ενδιαφέρει πολύ. Τους μόνιμους εισηγητές, προέδρους αντιπροσωπιών για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση είναι αφιερωμένη σε ένα ουσιαστικό σημείο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών και των μελών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν εφαντηρήσεων, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι ομιλητέ. Μάλλον, αγαπητοί ομιλητέ, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σασόλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ηγέτε των πολιτικών ομάδων, θέλουμε να ακούσουμε τι ιδέε έχετε. Πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάλαση, διάσταση μάλλον των μεταρρυθμίσεων εν ώψη ε, της διευρύνσεως, ομάδας εργασία Έχουμε τα μέλη που καλύπτουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Ραχοκοκαλιά της ομάδας είναι οι συγητές και οι πρόεδροι αντιπροσωπιών που ασχολούνται με τις χώρες της περιοχής σας. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Πάνω από 60% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέπετε είναι νεοεκλεγέντα μέλη. Εξελέγησαν το 2019 Οπότε αυτή είναι μια ευκαιρία να ρίξουμε μια φρέσκα ματιά. Λοιπόν, αυτή η σύνοδος κορυφής των Προέδρων είναι ένα βήμα προς πιο συντονισμένη, στρατηγική ε, και διευρυμένη συνομιλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ούτω ώστε να προωθήσουμε την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω ζητήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τη 24η Οκτωβρίου του 2019 όσον αφορά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Η Σύνοδος Κορυφής και η κοινή δήλωση είναι πρώτη στα παραδείγματα διπλωματίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε στιγμές όπου η διακυβερνητική διαδικασία δυστυχώς ε, έχει χάσει την ορμή της. Προτείνω λοιπόν να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση σαν μια μελλοντοστραφής συζήτηση μεταξύ εταίρων που έχουν παρόμοια προσέγγιση. Ε, οι εισαγωγικέ δηλώσεις ας κρατήσουν μόνο πέντε λεπτά και μετά ας προχωρήσουμε στην ουσιαστική συζήτηση που θα αφορά το μέλλον της διαδικασίας διεύρυνσης. Θα παρακαλούσα τους αξιότιμους συναδέλφους από τη Βοσνία Ζεγοβίνη να μοιραστούν ε, το χρόνο τους με ένα λεπτό παραπάνω ο καθένας. Θα είμαι αυστηρό και με του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ζητήσω την κατανόησή τους. Οι συγητέ και οι πρόεδροι της αντιπροσωπείας θα έχουν προτεραιότητα στη συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, αυτή την πρόταση που σας έκανα. Αυτό βλέπω. Συμφωνείτε. Καλό τους ε, ομιλητές να κάνουμε σύντομη εισαγωγή, να μας πείτε ποιο είναι το όραμά σας για την Ευρώπη και τη διεύρυνση και μπορείτε να απευθύνετε και ερωτήσεις προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Γκράμος Ρούτσι, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Αλβανίας. Σας ευχαριστώ. Είναι η τρίτη συνάντηση την οποία οργανώνουμε. Ε, είναι η πρώτη συνάντηση και προφανώ στην πρώτη συνάντηση σα παρουσίασα ποιο είναι το όραμά μα σε ό,τι αφορά την α, προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεύρυνση με τι χώρε μα. Εκ παραλίλου μίλησα και για το θέμα τη της απόφασης μη έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερη συνάντηση των επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων σας παρουσίασα τα αποτελέσματα τα οποία πέτυχε η χώρα μου σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αλβανία. Πρόκειται λοιπόν για την τρίτη υπαριθμόν συνάντηση. Προφανώς πάντα υπάρχει μία πρώτη φορά και αγαπητοί ευρωβουλευτές, αν ναι, οποιοδήποτε εδώ ερχόταν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο για να συζητήσουμε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Βεντικά Βαλκάνια, τις χώρες των Βεντικών Βαλκανίων. Αυτός αποτελούσε μεγάλη είδηση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Έχουμε άλλους πέντε συναδέλφους και έχουμε περάσει ώρες ολόκληρες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, τους εισηγητές και τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Όταν ε, είπα ότι πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά, αναφερόμουν στο γεγονός ότι δεν είμαι ενήμερος να υπάρχει στοιχεία προηγούμενο για συνάντηση με πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν γνωρίζω λοιπόν να υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση με τους εισηγητές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπεία για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό μας εντυπωσιάζει. Εντυπωσιάζει ιδιαίτερα και εμένα, να σας πω την αλήθεια, και πιστεύω ότι πρόκειται για μια νέα προσέγγιση, μια νέα εξέλιξη αν θέλετε. Μας δίνει λοιπόν ένα πράσινο φως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αποτελεί ενθάρρυνση. Μετά από την απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Για εμά, λοιπόν την Αλβανία και για την ε, Βόρεια Μακεδονία αλλά και για τις έξι χώρες που παρακολουθούν ΜΕΝ την πρόοδο των ΔΕ. Είμαστε λοιπόν έξι χώρε ε, σύνολο αλλά έχουμε τρεις διαφορετικούς ρυθμού αν θέλετε. Δύο έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσει, δύο άλλες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει την πραγματεύσεις και έχουμε και τους συναδέλφους από τη Βοσνία Ζεγοβίνη και τους ε, συναδέλφους από το 25 αντιμετωπίζουν περαιτέρω προβλήματα και δεν μπορούν καν να ωφεληθούν από το καθεστώς ελεύθερη μετακίνηση. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ε, και αυτή η συνάντηση αποτελεί κάτι το εξαιρετικά ενθαρρυντικό για μας. Το τελευταίο έτος ήταν δύσκολο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των νέων εξελίξεων. Αλλά και λόγω των ευρωεκλογών που διοργανώθηκαν. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων ακολούθησαν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ από ό,τι και οι ίδιοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα Μα είχαν προειδοποιήσει ότι πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη άνοδο των ευρωσκεπτικιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είπα ότι είμαι εντυπωσιασμένο. Με έχει εντυπωσιάσει το γεγονό ότι είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Διεύρυνση δίνει σύσταση για έναρξη διαπραγματεύσεων. Δύο φορέ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσταται. Δεν ξέρω να έχει υπάρξει άλλη τέτοια απόφαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι υπάρχει νέο κοινοβούλιο, 65% των μελών του κοινοβουλίου είναι ουσιαστικά νέοι βουλευτέ. Μα εντυπωσιάζει λοιπόν το γεγονό ότι οι βουλευτέ αξιολόγησαν τη διαδικασία αυτή και την έκριναν άδικη. Αυτό πραγματικά μα ενθαρρύνει ω πολιτικού και μιλώ τώρα εξ ονόματο τη Αλ Αλβανία και για του συναδέλφου από την Βόρεια Μακεδονία που έχουν την ίδια άποψη. Και θα ήταν πραγματικά πολύ καλό στην επόμενη σύνοδο να διορθωθούν αυτά που έγιναν λάθος στο παρελθόν. Και ελπίζουμε λοιπόν να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Είμαι λοιπόν ε, πεπισμένος και αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα ληφθεί η απόφαση αυτή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω και να σα ευχαριστήσω για την ε, παρέμβασή σα. Ευχαριστούμε και εμεί για την παρέμβασή σα και τώρα να πάρει το λόγο ο κύριο Ντενίς Σβίτζετ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων από τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ήμουν εδώ παλιά, εδώ και κάποια χρόνια. Σε κάποιο συμβούλιο, κάποια συνεδρίαση που είχαμε, χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εθνοσυνέλευσης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις για θέματα οικονομικά και ασφαλείας. Στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, τη Βοσνία Αρσεγοβίνη. Κυρίως εν ώψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους από άλλα κοινοβούλια της περιοχής μας. Από τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι νοτιοδυτική Ευρώπη η περιοχή μας. Γεωγραφικά και πολιτικά ανήκουμε στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας Εζεγοβίνης και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορώ να μιλήσω εμπεριστατωμένα για τα προβλήματα της Βοσνίας Εζεγοβίνης καθώς και για ενδεχόμενες λύσεις που θα πετάχυναν τη διαδρομή της Βοσνίας Εζεγοβίνης προς το να γίνει μέλος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και να εξασφαλιστεί έτσι ειρήνη και ευημερία για τη χώρα. Το 2016, 2017 και 2018 ήταν δύσκολα χρόνια για τη Βοσνία Ζεγοβίνη όσον αφορά την ένταξή της. Όμως κάναμε προσπάθειες με ενθουσιασμό. Παρά τις δύσκολες πολιτικές περιστάσεις, διατηρήσαμε τη σταθερότητα, αναπτυχθήκαμε οικονομικά, διαφυλάξαμε ε, την ανεξιθρησκεία που είναι η μάγνα κάρτα της ύπαρξής μας. Έχουμε μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια αξία που θα φέρει, θα συνεισφέρει με αυτήν, με την ιστορία μας η Βοσνία Ζεγοβίνη, στον πλούτο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε να συμφιλειωθούμε με τους γείτονές μας και θέλουμε να σεβόμαστε και την κυριαρχία των άλλων χωρών. Η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν είναι μεγάλη χώρα. 3,5 εκατομμύρια κατοίκου έχουμε μόνο. Αλλά είχαμε πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστε πέρσι. Είχαμε αύξηση το ΑΕΠ πάνω από 3%. Υγούμεθα στι εξαγωγέ στην περιοχή. Και είμαστε στι πρώτε 10 χώρες όσον αφορά τις εξαγωγές. Οι 7 άλλες χώρες είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν έχουμε εναλλακτική από την ένταξή μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κατάλληλες υποδομές, να δημιουργήσουμε κοινωνία της γνώσης. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική μας ανάπτυξη. Θέλουμε καλύτερες προδιαγραφές και ειρηνική ζωή για τους, νέους πολίτες, για τους πολίτες μας μάλλον. Αλλιώς θα εξακολουθούν να φεύγουν οι νέοι. Και όλα αυτά που συζητούμε σήμερα δεν θα έχουν νόημα αν φύγουν οι νέοι. Θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους στην περιοχή, διότι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την περιοχή μας. Θέλουμε ενοποίηση της χώρας, να υπάρχει η προοπτική α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πλήρους ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξαλείψουμε τις αρνητικές πτυχές. Όλα αυτά που οδήγησαν στον πόλεμο της δεκαετίας του 90. Θέλουμε να ανοιχτούμε προς το μέλλον, να δεχτούμε τις ευρωπαϊκές αξίες, να υπάρχει θετική πολιτική βούληση, να έχουμε συνένεση όχι μόνο στα λόγια, να ενστερνιστούμε τις ευρωπαϊκές αρχές, να αλλάξουμε την δική μας ένωμη τάξη και να μπορούμε να σωματώσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο γρήγορα στην ένωμη τάξη μας και έτσι η Βοσνία Ζεγοβίνη να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό με τις ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, εμείς τη Βοσνία Ζεγοβίνη δεν θέλουμε προνομιούχα σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να μπούμε σε κάποια ε, πρωτοβουλία περιφερειακή που θα αντικαθιστά την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να γίνουμε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι πολύ σοβαρό έργο αυτό, δύσκολο καθήκον, αλλά για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Βοσνίας αζεγοβινης για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας καλούμε να μας βοηθήσετε να μπούμε στην επόμενη φάση της ένταξης της Βοσνίας αζεγοβινης Να προχωρήσουμε φέτος, να αποκτήσουμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας φέτος. Σας καλούμε να το κάνετε αυτό όλοι μαζί να κινηθούμε και έτσι η Βοσνία Ζεγοβίνη να μπορεί να διαφυλάξει την ειρήνη, τη σταθερότητα και να είναι πολυπολιτισμική χώρα, να συνεχίσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη και την περιφερειακή συμφιλίωση. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πίτσουλα, στον κύριο Ντραγκάντσοβιτς τώρα, που είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βοσνίας Εζεγοβίνης. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, κυρίοι βουλευτές. Μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα να ε, κάνω και εγώ μια εισήγηση μετά από τα όσα είπε ο κ. Έχουμε συνένεση όσον αφορά την ιδέα ότι η Βοσνία πρέπει να προχωρήσει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε εναλλακτική. Θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι ο χρόνος που χάθηκε τον την περασμένο έτος ε, χαρακτηρίστηκε από κοινέ προκλήσεις. Χρειάστηκε να ασχοληθούμε με την επίλυση ορισμένων εσωτερικών προβλημάτων, αλλά στη διάρκεια των τελευταίων δύο-τριών μηνών ανοίγεται νέα προοπτική στα διάφορα διοικητικά κλιμάτια και θεσμικά κλιμάκια της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και είναι αναγνωρίσιμη μία νέα ορμή που στόχο έχει να λύσει τι ε, προβλήματα και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που μας ε, καθυστέρησαν μέχρι τώρα. Πρόκειται για την, ε, τον εκλογικό νόμο ε, που ε, καθορίστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από το, της Βοσνίας αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα όσα μας εμποδίζουν να μπορέσουμε λοιπόν να τα ανακαλέσουμε. Μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό να τα ανακαλέσουμε όλα αυτά άμεσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε μέχρι το Μάρτιο να μπορέσουμε να τα μεταρρυθμίσουμε με την εκλογική μας νομοθεσία. Είναι ένα ζήτημα επί το οποίο εργαζόμαστε εδώ και χρόνια ε, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην Προεδρία της χώρας, ώστε να εκπροσωπούνται σωστά οι τρεις ε, ε, λαοί που ζουν στη χώρα μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις παρεξηγήσεις που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να φροντίσουμε ώστε οι θεσμοί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να εφαρμόσουν ε, προδιαγραφές ευρωπαϊκού επίπεδου που ισχύουν σε όλα τα κράτη δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι η θα πρέπει να έχουμε ελευθερία τύπου, αλλά και όλα όσα είναι απαραίτητα για την οικονομία της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ε, θέλουμε δε να πετύχουμε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ούριο άνεμο, και με ρεαλιστικές προθεσμίες να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες εργασίες ε, πριν τη διάσκεψη κορυφής του Μαΐου τη διάρκεια της οποίας αναμένονται δηλώσεις όσον αφορά τη στρατηγική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διεύνηση διάσκεψη κορυφής όπου θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δοθεί σαφής προοπτική στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Φυσικά με τη δική σας ε, ε, ε, στήριξη μπορούμε να το καταφέρουμε γιατί υπάρχουν μόνο δύο πιθανότητες. Από τη μια πλευρά η ολοκλήρωση και από την άλλη η είναι η εγκατάλειψη αυτής της ε, προπτικής. Εγώ ελπίζω πως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά μέχρι τότε ώστε να έχουμε τη δική σας ενθάρρυνση ως υποψήφια χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόγιουφτσα, πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κωσυφοπεδίου. Τώρα. Μούγκα. dhe takime Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνάντηση. Αν με ακούτε, με ακούτε, πολύ ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Πιτσουλά και τους ευρωβουλευτές. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο φιλικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ενοποίησης των Δυτικών Βαλκανίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ιδιαίτερως τη διοργάνωση της δραστηριότητα αυτής από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή των ε, Προέδρων των Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων. Οι πιο πολλές χώρες της περιοχής έρχονται από κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε. Και είμαστε στο επίκεντρο λοιπόν των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στι εκάστοτε χώρε μα. Οι κοινοβουλευτικέ ε, συναντρήσει, συνελεύσει. Ασχολούνται με την νομοθεσία που έχει ως σκοπό την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ασχολούμαστε με το έργο της κυβέρνησης που στο σκοπό έχει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αποτελούν ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και καθορίζουν και την ταχύτητα της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε ψευδέστηση. για τη μεταρρύθμιση και την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υπάρχουν κοινοβούλια τέτοιου τύπου στι χώρε μα Και υπό την έννοια αυτή, ακόμα και η διοργάνωση τη εκδήλωση αυτή, η οποία έχει ω σκοπό την ενδυνάμωση, ακριβώ, την ενίσχυση των ε, κοινοβουλίων, είναι πραγματικά κάτι το οποίο χρειάζεται αν θέλουμε να κάνουμε σταθρά βήματα προς την ενοποίηση, λαμβάνοντα υπόψη και τα διάφορα επίπεδα της ενοποίησης, το κοσυφοπαίδιο είναι το τελευταίο. Το τελευταίο στη λίστα των χωρών των βεδικών Βαλκανίων. Είμαστε λοιπόν στη φάση υλοποίησης και εφαρμογής της Συμφωνίας ε, Σταθεροποίησης. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξή. Τα τελευταία χρόνια λόγω της χαμηλότερης ταχύτητας των πολιτικών διαδικασιών και λόγω των μέτρων που είχαμε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σταθεροποίησης, μόνο 50 έως 60% των μέτρων αυτών τελικά υλοποιήθηκαν, εφαρμόστηκαν. Από την άλλη αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς ότι αυτές οι ιστορικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται και με τις εκτορικές διαδικασίες. Υπάρχει λοιπόν μια διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο διαστάσεων και συχνά εξαγάγουμε διδάγματα από αυτά που συνέβησαν στην γειτονική μας χώρα, την Νότια Μακεδονία, που όπως ξέρετε έχει υλοποιήσει τη διαδικασία αυτή. Το 2005, 14 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, για να περάσουν δηλαδή από το ένα βήμα στο επόμενο την εκκίνηση, την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό λοιπόν και η μελλοντική κυβέρνηση είναι πλήρως προετοιμασμένη προκειμένου και η διάσταση αυτή η εξωτερική και οι καλές γειτονικέ σχέσεις, οι καλές σχέσεις γειτονία με τις ε, όμορες χώρες να μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση ακριβώς αυτή της ε, υπέρβασης των εμποδίων και το πέρασμα στην επόμενη φάση τη διαδικασία. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την σημερινή εκδήλωση και ενδεχομένω να γνωμοδοτήσουμε και λίγο πιο μετά, να τοποθετηθούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρο, για την ε, παρέμβασή σα. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ιβαν Μπράμπιτ από το Μαυροβούνιο. Σα ευχαριστώ. Αυτό ο διάλογο με του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πραγματικά χαρά για μένα. Πρέπει να πω ότι διαπιστώνω ότι ακόμα και οι βουλευτές που ήδη ε, εκτελούν τη θητεία αυτή, την πιο μακρά θητεία στο Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσαν ότι ήταν η πρώτη φορά που προσεκλήθημεν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Αν γινόταν περισσότερε τέτοιε συναντήσει κατά το παρελθόν, θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στι διευρύνσει και ίσως θα υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ανεξάρτητα από αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνοδο κορυφής και ευχαριστούμε πολύ που σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκδηλώσατε τη διαφωνία σας με την τροχοπέδη που ετέθη στη διαδικασία διεύρυνσης. Όπως πάντα, όταν βλέπουμε αρνητικά γεγονότα, προσπαθώ να βρω τις θετικές πτυχές. Και αν κάποιοι, ε, κάποιες χώρες δεν θέλησαν να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, αυτό επηρεάζει την περιοχή τη δική μας, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ξανά όμως από αυτό το γεγονός συγκεντρώθηκαν οι προβολείς επάνω μας. Ειδού, εξ αυτού έχουμε και αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ και νέο τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ επίση για την έξοχη ανταλλαγή απόψεων τη περασμένη εβδομάδα στην Ποντγκορίτσα, όταν ο κ. Πιτσούλα για πρώτη φορά ο πρόεδρος πήγε για πρώτη φορά, ήρθε πρώτη φορά σε εμά. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχετε καλή κατανόηση του διακυβεύματος για την περιοχή. Και έτσι έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχιστεί η διαδικασία. Αυτή η συνεδρίαση τώρα, αυτή η συνάντηση με τους προέδρους, συμπροέδρους, όχι μόνο των κοινοβουλίων, αλλά και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, των καθήλια αρμοδίων, κυρίω τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι επιφορτισμένη με τη διεύρυνση, αυτέ οι συναντήσει είναι μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε εκ νέου την ανάγκη να αποστείλουμε σαφέ μήνυμα υπέρ τη διευρύνσεω προ την Ευρώπη την Νοτιοανατολική. Τέθηκε μια ημερομηνία η 5η Φεβρουαρίου. Ε, συζητήσαμε με τον Επίτροπο των Αρμόδιων για τη Διεύρυνση χτες στις Βρυξέλλες μου επιβεβαίωσαν ότι Μαυροβούνιο και η Σερβία προχωρούν στις διαπραγματεύσεις και θα είναι και πιο ορατά τα αποτελέσματα. Τι θα γίνει όμως με τις χώρες εκείνες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διαπραγματεύσεις. Πάντως θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ στους γείτονές μας τη Σλοβενία και την Κροατία ε, ότι πάντα μας υποστήριζαν. Πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα τι περιμένουμε μένα από τους δε. Να καθορίσουμε κριτήρια και τους πύχες που θα θέσουμε τη διαδικασία και ποιοι θα είναι οι ρόλοι δικοί μας που θα παίξουμε στην όλη διαδικασία της ένταξης, τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε και τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινό καθήκον είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα αυτής, να έχουν πάλι εμπιστοσύνη οι πολίτες. Αντιμετωπίζει προβλήματα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Αυτό δεν αποκλεί όμως επουδενή τη διεύρυνση. Χρειάζεται να προχωρήσουμε όλοι χέρι με χέρι για να απαγιωθεί αυτή η διεύρυνση. Οι πολίτε του Μαυροβουνίου επιθυμούν σαφήνεια, ορατότητα όσον αφορά τη διαδικασία διεύρυνση και να συνεχιστεί αυτή. Ίσως να διαφέρουν δικές μας θέσεις από τις άλλες χώρες της περιοχής, ίσως γιατί εμείς θα είμαστε πιο προχωρημένοι όσον αφορά τη διαδικασία. Μη λησμονούμε όμως ότι εδώ και 8 χρόνια είμαστε, συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω, όπως και άλλοι, ότι το μονοπάτι είναι εξίσου, η διαδρομή είναι εξίσου σημαντική όπως ο τελικός σκοπός, δηλαδή η προσχώρηση. Βέβαια από τη στιγμή που το μονοπάτι δεν είναι πάρα πολύ μακρύ. Το 2025 ήταν η πιο κοντινή προπτική που θέσατε για ένταξη, ίσως πιο αργά για τη Σερβία. Φανταστείτε ποια θα είναι η προθεσμία για την Αλβανία ε, και τη Βόλια Μακεδονία και ποια θα είναι η ημερομηνία για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Υπάρχει ασάφεια εκεί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία. Η περίοδος αβεβαιότητας, κρίσης και προβλημάτων πρέπει να μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε αποφασιστικά χωρίς να αλλάξουμε τα θεμέλια της διαδικασίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό εγχείρημα με τα πολεμικά και η διεύρυνση σίγουρα είναι η σημαντικότερη πολιτική της Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20 διότι είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διπλασιάζεται τον αριθμό των κρατών μελών της. Κάποια μέρα ελπίζουμε όλα τα κράτη-μέλη των Δυτικών Βαλκανίων να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να ενταχθούν η κάθε χώρα σύμφωνα με την αξία της. Να κριθεί κάθε χώρα ανάλογα με τα επιτεύγματά της και τη θέση της. Δεν πρέπει να αρκούμε απλά μηνύματα που θα αποστέλλονται στον αφορά τη σημασία της διεύρυνσης, της συμφιλίωσης και της εργασίας. Είναι σημαντικό απτά αποτελέσματα να γίνονται αισθητά και να γίνουν αισθητά γρήγορα. Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου εργάζεται ε, πυρετοδός για αυτό το σκοπό, ενισχύει τον υποπτικό έλεγχο όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσία. Κατά 40% έχουμε ολοκληρώσει τι διαβουλεύσει επ' αυτού, κυρίω πέρσι. Θα κινηθούμε υπέρ των νέων και υπέρ τη κοινωνία των πολιτών και θέλουμε να ξέρουμε τι εμπειρίε έχετε σε αυτό όσον αφορά τη συνεργασία με χώρε περιοχή. Διοργανώνουμε πολυάριθμε διασκέψει και συνέδρια και το κοινοβουλευτικό φόρουμ ε, που διοργανώνεται εδώ και 16 χρόνια που διοργανώνουμε είναι μια καλή βάση για συνεργασία περιφερειακή των κοινοβουλίων. Ευχαριστώ και πάλι. Εσείς πιστεύω οι ίδιοι που είσαστε εισηγητέ ή συμπρόεδροι και στις Βρυξέλλες και στις διάφορες χώρες σας παίζετε το σημαντικότερο ρόλο και θα ήθελα να σας ζητήσω, να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε ε, ακόμα περισσότερο το κοινό εγχείρημα της ΕΕ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τώρα τον κύριο Τζαφέρη, τον πρόεδρο της συνεδρεύσεως της Βορείου Μακεδονίας να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους εισηγητές και τους συμπροέδρους. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ειδωθούμε, να συζητήσουμε ζητήματα που μας προβληματίζουν. όσον αφορά την επίτευξη του απότερου στόχου μας, δηλαδή της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προχωρήσει πολύ από τότε που συνήθη η Συμφωνία ε, Σταθεροποίησης και από τότε που υποβάλαμε αίτηση ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα χρόνο αργότερα δε επιτύχαμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Το 2009, μετά από τέσσερα χρόνια δηλαδή, είχαμε την πρώτη θετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πράγμα που συνοδεύθηκε από την απόφαση του απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της χώρας μας. Έκτοτε, μέχρι και πέρυσι, είχαμε 10 θετικές εκθέσεις και 10 συστάσεις για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν και οι προσδοκίες μας. γιατί λάβαμε υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο που είχαμε επιτύχει. Είχαμε σαφή σύσταση τον ε, Ιούνιο. Ε, περάσαμε την απογοήτευση του Οκτωβρίου όταν δεν εγκρίθηκε η απόφαση για την ανέξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, επιμένουμε. Το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο πέρυσι, που έδωσε πλήρη στήριξη στις χώρες της περιοχής, είναι ένα φως στην άκρη του τούνελ που, ε, για την ώρα. Και ελπίζουμε πως αυτή τη φορά θα εγκριθεί και η νέα μεθοδολογία διεύρυνσης και η απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις ε, χώρες ε, τις γειτονικές μας. Ελπίζουμε πως θα προχωρήσουν όλα παράλληλα και ότι η απογοητευτική απόφαση του περασμένου Οκτωβρίου χρησιμοποιήθηκε από τους ε, πολιτικούς ηγέτες ως ένας τρόπος για υιοθέτηση απόφασης για την ε, διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Ξέρετε ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές στις 12 Απριλίου και ότι με αυτές τις ε, εκλογές θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και πάλι την στήριξη για να συνεχίσουμε στον ευρωπαϊκό μας, στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Ελπίζουμε πως οι εκλογές θα οργανωθούν όπως αναμένεται, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες από το 2016 οργανώθηκαν από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και ο κύριος ρόλος αυτής της κυβέρνησης ήταν να οργανώσει ε, ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές. Τον Ιανουάριο λοιπόν ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακή κυβέρνηση και έχουμε και ημερομηνία για την ε, διάλυση του Κοινοβουλίου, οπότε θα αρχίσει και η προεκλογική περίοδος. Έχουμε τη διαδικασία του Ζαμονέ, έχουμε τη διαδικασία του Βερολίνου και ελπίζουμε πως η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2022 θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε ενεργά και να μπορέσουμε να ε, ε, παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για το ευρωπαϊκό μέλλον στην ε, συνέλευση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και αν έχετε ερωτήσεις ευχαρίστω να τις απαντήσω. Να καλέσω λοιπόν τώρα την κυρία Μάγια Βοϊκοβίτς να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιτσουλακή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου τους ε, πρόεδρους των κοινοβουλίων των Βετικών Βαλκανίων που πήραν το λόγο πριν από μένα. Οι συνάδελφοί μου προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν ως χώρες που προσπαθούν, καταβάλουν προσπάθειες και αγωνίζονται να γίνουν σε κάποια φάση μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια στιγμή. ε, το χρονόμετρο δείχνει ότι έχω ήδη μιλήσει 6 λεπτά. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει νόημα λοιπόν να συνεχίσουν να επαναλαμβάνω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι μελητέ. Είσαστε εισηγητέ ε, εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι χώρε μα. Και θα ξέρετε λίγο πολύ τα πάντα για τις χώρες μας, για τις πολιτικές μας φιλοδοξίες και για τις ε, εσωτερικές πολιτικές μας και για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, στις χώρες μας. Δεν έχει νόημα λοιπόν να παρουσιάσω τον εαυτό μου και τη χώρα μου στα μέλη της Επιτροπής της Αντιπροσωπείας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό θα σήμαινε προβλήματα. Δεν είμαστε ο μεγάλος άγνωστος για σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω πραγματικά να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε να μιλήσουμε ανεκτά εδώ στις Βρυξέλλες για την πολιτική διεύρυνση και κυρίως ότι αφορά τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια ή την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως το θέλετε το λέτε. Και είμαι περήφανη που εκπροσωπώ μια χώρα από αυτό το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επίρου. Αυτό που έχω να σχολιάσω εγώ είμαι για πρώτη φορά στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητάμε για το κατά πόσον και εφόσον η Σερβία κάποια στιγμή θα είχε τη δυνατότητα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι για δεύτερη θητεία πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου και για πρώτη φορά έρχομαι εδώ για να συζητήσω τη μοίρα της χώρας μου ως ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και αυτός ήταν ο κατεξοχήν ο, ο πρώτος και πιο σημαντικός ε, στόχος μας στην εξωτερική μας πολιτική. Να είμαστε εδώ. Είχαμε μία συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνυπογράψαμε μία δήλωση που αποτελεί ένα μικρό δείγμα εμπιστοσύνη προς όλους μας. Γιατί όλοι μείναμε έκπληκτοι και έχουμε... Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε με την απόφαση να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με την ε, Βορειομακεδονία και την Αλβανία. Και πρέπει να πω ότι αυτό ήταν πραγματικά πολύ αρνητικό μήνυμα το οποίο εστάλει όχι μόνο προς τους πολίτες των δύο χωρών, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω λοιπόν αυτή η συνάντηση και η συνομιλία μαζί μας να μην αποτελέσει κάτι το μεμονωμένο και να υπάρξει συνέχεια. Ελπίζω το Κοινοβούλιο λοιπόν να το πάρει αυτό στο σοβαράκι, να κινηθεί η Ένωση πέρα από το δίλημα αυτό για το κατά πόσο θα αρχίσουν ή δεν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Η Γαλλία ήταν μοναδική η οποία μίλησε ανοιχτά, αλλά Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το δίλημα για τον κατά πόσο θα υπάρξει διεύρυνση ή όχι είναι ένα ερώτημα το οποίο πλανάται ή και είναι κρεμές. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε την Ένωση να ξεπεράσει το φόβο για το πόλητες των Δυτικών Βαλκανίων, και είμαστε κάτι φρικτό, το οποίο είναι κάπου στον ορίζοντα και το οποίο θα χτυπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπάντεχα αν ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων ε, εφόσον φυσικά διαπραγματεύσει ή αν υπάρξει επιτάχνηση των διαπραγματεύσεων εφόσον φυσικά εκπληρωθούν οι όροι. Τι είναι λοιπόν αυτό το φριχτό που φοβάται η Ευρώπη. Τι μελιγενέστε αν αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Αναμέναμε η ευρωπη τι λιγινέστε αν λοιπόν υποστηρίξη Πήραμε αυτή την υποστήριξη λοιπόν και πάλι. Είμαστε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε με πάσα ειλικρίνεια να μην είναι το τέλο αυτό τη διαδικασία αυτή, να είναι μια και μοναδική εμφάνιση αυτή. Θέλουμε να είμαστε τέρι στη διαδικασία αυτή και πείτε μα λοιπόν πώ μπορούμε να βοηθήσουμε και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει τον φόβο αυτό και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει. η... για το κατά πόσο λοιπόν θα παραμείνει κλειστή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Υπάρχει λοιπόν καλή εκπροσώπηση και καλά κοινοβούλια. Ακολουθούμε τα ορόσουμε και να αρμονιζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχουμε καλή συνεργασία σε επίπεδο ένας προς ένας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Θα θέλαμε από πλευρά μα να μην συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο όταν υπάρχουν θέματα τα οποία θεωρείται ότι είναι προβληματικά από πλευρά μα. Θα θέλαμε αυτή η συνεργασία να είναι ένα αμφίδρομο, ανοιχτό κανάλι. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, τους προέδρους για αυτά τα εισαγωγικά σχόλια. Τώρα ήρθε η ώρα των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Καταρχάς, στους εισηγητές και στους προέδρους αντιπροσωπείων θα ήθελα να δώσω το λόγο. Αλφαβητικά, και τρία λεπτά ο καθένα, παρακαλώ το πολύ. Όσο μπορούμε να το τηρήσουμε αυτό. Για να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Πρώτος, Ισαμπέλ Σάντο. μόνιμη συγγήτρια για την Αλβανία. Ισαμπέλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους προέδρους των Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων που είναι σήμερα παρόντες. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή. Είναι μια στιγμή όπου το Ευρωκοινοβούλιο, εμείς οι θεμητοί, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λαών μας, των ευρωπαϊκών λαών, αναλαμβάνουμε μια δέσμευση μαζί σας. Μια δέσμευση που εμείς ε, έχουμε ε, ε, εξάλλου ε, ήδη αφήσει έντυπη στο ψήφισμα που ήδη έχουμε εγκρίνει πριν από λίγους μήνες. Ο λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης θα μείνει πιστή αυτός ε, μέχρι το τέλος. Και ακριβώς αυτή είναι η δέσμευση ε, που ανέλαβαν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια και όλοι όσοι συνυπέγραψαν δηλαδή το ψήφισμα, υπερψήφισαν το ψήφισμα, ε, διατηρούμε τη δέσμευσή μας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Είπαμε ότι πρόκειται για μία πρώτη συνεδρίαση, ελπίζω πως θα είναι η πρώτη από πολλές συνεδριάσεις τέτοιε που θα κάνουμε μεταξύ μας, έτσι ώστε ανάμεσα στα διάφορα κοινοβούλια να διατηρήσουμε μία μόνιμη επαφή, μία μόνιμη συνεργασία και έναν μόνιμο διάλογο με στόχο να προετοιμάσουμε καλύτερα τη διαδικασία, την πρωτοεξιακή για κάθε χώρα γιατί ακριβώς ε, τα κοινοβούλια θα συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες μέσω των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν και θα έχουν ε, πολύ κύριο ρόλο, λιώδη ρόλο να παίξουν τα κοινοβούλια των χωρών σας. Ε, μέχρι τέλους, το μόνο που εγώ θέλω να ζητήσω είναι ότι η λιγότερη ευτυχή στιγμή εκείνη του Οκτωβρίου στο Συμβούλιο θα μείνει μόνο αυτό, μια στιγμή ατυχής και ότι στις χώρες σας, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα συνεχίσετε τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές όχι μόνο επειδή ε, ε, από αυτό εξαρτάται η πρωτεξιακή πορεία των χωρών, αλλά είναι σημαντικές ούτως ή άλλως για την ε, δημοκρατία στις χώρες σας και για την καθημερινή ζωή των πολιτών σας. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει καθόλου να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Θα σε ενθαρρύνω θερμά να συνεχίσετε με την ίδια ταχύτητα και από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να βασίζεστε στη δέσμευσή μας, στην προσήλωσή μας, στην διαδικασία αυτή μέχρι τέλους είναι προφανές πως υπάρχει σημαντικός υπερβολικός μάλλον ε, γραφειοκρατικός φόρτος, ότι η διαδικασία πρέπει να αναθεωρηθεί. Ναι, συμφωνώ και εγώ, πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει όλος, όλη η πορεία που έχει γίνει μέχρι τώρα να συνεχίσει και να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, χωρίς καθυστερήσεις ε, και πάυσεις ε, Και όπως είπα, εμείς παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, πρόεδρος αντιπροσωπείας για την Αλβανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την έναξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία εκφράζει βαθιά απογοήτευση όσον αφορά την αποτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες αυτές χώρες. Η Αλβανία από όταν τη δόθηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας τον Ιούνιο του 2014 είχε κάνει αποφασιστική πρόοδο για την εκπλήρωση των στόχων των σχετικών με τις πέντε βασικές προτεραιότητες για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Απ' την άλλη πλευρά, η αλβανική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερο τα παρόντα προβλήματα. Πραγματικά παραμένω αισιόδοξο και πιστεύω ένθερμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει σε συνένεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την διεύρυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βιόλα Φων Κρεμόν Τάουμπερ, που είναι μόνιμη εισηγήτρια για το Κωσφό Πέδιο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι. Πραγματικά είμαι, έχω εντυπωσιαστεί, διότι αυτό που έχετε κοινό είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που τηρήσατε, τα τεχνικά κριτήρια που τα περισσότερα έχετε πληρώσει είτε για απελευθέρωση των θεωρήσεων όπως το κοσυφοπαίδιο ε, είτε για τις συνομιλίες τις ενταξιακές. Σε αυτή τη φάση κατανοώ ότι η ατμόσφαιρα και η διάθεση στις χώρες σας δεν είναι αισιόδοξη, δεν είναι θετική. Ε, Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ πάρα πολύ τη συνεργασία σας, ότι είστε ανοιχτοί, ότι εμφανιστήκατε, ότι είσαστε έτοιμοι να παραμείνετε σε ένα πλαίσιο καλής σταθερής συνεργασίας. Το εκτιμούμε πολύ εμείς εδώ που παριστάμεθα. Βέβαια, όπως και άλλοι τόνισαν, είναι σωστό να μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας, σε εμά τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, διότι σας υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε την διεύρυνση. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σίγουρα είναι υπέρ αυτής και έχουμε διάφορα ψηφίσματα που αυτό ακριβώς τονίζουν. Είπε η κυρία Πρόεδρος και ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε. Και κάποια από εσά αναφερθήκατε στις επικείμενες εκλογές. Κάποια από εσά έχετε μόλις βγει από εκλογές και περιμένουμε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το να είναι σταθερή περιοχή θα ήταν κάτι καλό το είπε και η Ζαμπέλ για να τονωθεί η μεταρρύθμιση εσωτερική σε όλους τους τομείς, ούτως ώστε στους πολίτες να δώσετε αυτά που περιμένουν. Παραδείγματος χάρη μια κυβέρνηση, αλλά και ποιοτική υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση. Όλα αυτά θα μας δώσουν το συνέστημα ότι δεν προέρχεται εκ των έξω κατόπιν πιέσεως, αλλά ότι είναι εσωτερικό το κίνητρό σας και η φιλοδοξία σας να βελτιώσετε την κατάσταση των χωρών σας. Δηλαδή από τη μία ελπίζουμε ότι δίνουμε χρήματα, δίνουμε εργαλεία και εσείς από την άλλη τελικά εφαρμόζετε τα αναγκαία ούτω ώστε οι πολίτες σας να ζουν καλύτερα από ό,τι πριν. Όσον αφορά τον πλουραλισμό, τον πολυκομματισμό, το λέω στρεφόμενοι προς τη Σερβία, θα ήταν σημαντικότατο μήνυμα αν η αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα να μπορούσε να συμμετάσχει. Και το πολιτικό πλαίσιο σε αυτή τη χώρα να μην έχει την εξωφρενική μορφή που έχει τώρα. Εγώ θα έλεγα αν συνεχίσετε με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και πραγματικά εφαρμόσετε ποικιλομορφία κομματική και επιδιώξετε την εφαρμογή δημοκρατικών θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους υποψήφιους των επικειμένων εκλογών, για μας τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την επίσκεψη του ΗΠΑ του εκπροσώπου που θα γίνει η Πέμπτη και Παρασκευή θα θεωρήσουμε ότι γίνεται σημαντικό βήμα στην ε, περιοχή. Ευχαριστώ. Βιόλα Φρον Βλάντιμιρ πρόεδρος, αντιπροσωπεία συμπρόεδρος για το Μαυροβούνιο. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ε, κυρία Πρόεδρο και όλους τους κυρίους ε, πρόεδρους. Και πραγματικά είναι μοναδική αυτή η ευκαιρία. Ελπίζω ασφαλώς να μην είναι μία και μοναδική αυτή η ευκαιρία που έχουμε. Χρειάζεται ένα διάλογο και μάλιστα τακτικά, συχνά. Εδώ, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και στις χώρες σας, στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να υπάρξει λοιπόν ένας ε, πραγματικός διάλογος. Αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, σε θεσμικά όργανα φιλικά προς τη διεύρυνση. Χρειαζόμαστε όμως και πολλούς φίλους για τη διεύρυνση. Να υπάρξει πραγματικά πολιτική όθηση και ορμή σε κάποια χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνοδος λοιπόν αυτή δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά θεωρώ ότι αποστέλλει και ένα πολιτικό μήνυμα. Ελπίζω να επηρεάσει και τις ε, και άλλες υπηρεσίες και τα άλλα θεσμικά όργανα, την Επιτροπή και τα άλλα κρατημέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ και να συμφωνήσουμε και επί της ουσίας τι είναι αυτό που συζητάμε σήμερα και τι σαφή μηνύματα θα πρέπει να προωθηθούν σε όλη την περιοχή, στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη στη διεύρυνση και προφανώς χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη από πλευρά σα για τις υποσχέσεις μας. Δεν ε, μπορούμε να έχουμε άλλα διστακτικά μηνύματα όπως αυτό του Οκτωβρίου του περσινού έτους. Ελπίζουμε λοιπόν να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τις εναρξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και την Βόρειο Μακεδονία. Το νωρίτερο θα ήταν ο Μάρτιος του φετινού έτους. Αυτό θα ήταν υπέροχο μήνυμα για όλη την περιοχή γιατί θα έχουμε και σημαντικό έτος εκλογών στην περιοχή και στο Μαυροβούνιο ε, περιμένουμε εκλογές στο φθινόπωρο αλλά και στη Βόρεια Μακεδονία πιο πριν και στη Σερβία ασφαλώς. Η συνάδελφος ε, είπε πόσο σημαντικές ήταν είναι αυτές οι εκλογές για την ε, διάσταση την ευρωπαϊκή. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το μήνυμα. Θα ήθελα να τονίσω ένα στοιχείο, την ελευθερία έκφρασης και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Εξαιρετικά σημαντικά αυτά σε ό,τι αφορά μια σωστή δημοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενεργά κοινοβούλια. Και το λέω αυτό ως ένα άτομο που σχολιάζει και την δολοφονία δημοσιογράφου ερευνητικής πριν από δύο χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν να αναφερθεί αυτό και στη Συνοδό για το μέλλον της Ευρώπης και προσβλέπω σε οποιαδήποτε συνάντηση περαιτέρω μαζί σας γιατί πιστεύω σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ελχάν Κιουτσούκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτσουλα. Κυρίε και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλώ ενώπιόν σας. Δεν βλέπω να υπάρχουν δύο πλευρές, γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη διεύρυνση είναι περίπλοκος. Θέλω να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση. Για μας λοιπόν ο αντικειμενικό στόχο είναι πώ η διαδικασία διαβρύνση μπορεί να γίνει πιο απτή, πιο ανοιχτή και να προσανατολιστεί πιο συγκεκριμένα σε αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια πλευρά του θέματο. Κοιτώντα όμω ε, και τις τελευταίες έρευνες από το Ευρωβαρόμετρο αναφέρουν ότι 67% των Αυστριακών δεν είναι υπέρ της διαβρύνσης. 64% των Γερμανών, και 63% των Γάλλων δεν είναι υπέρ τη διεύρυνσης. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε μαζί. Πώ μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη και την εντροπία που επικρατεί στις κοινωνίε αυτέ. Αυτό είναι δουλειά για όλου μα. Και πιο σημαντικό θεωρώ είναι το εξή. Μέχρι την διάσκεψη του Ζάγκρεπ, ακόμα και πιο πριν, Πώ μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις πολιτικές ανάγκες και τις πολιτικές αποφάσεις που θα λάβουν αυτές οι χώρες. Γιατί να θυμόμαστε τι συνέβη και τον Οκτώβριο του περσινού έτους. Όχι μόνο για να επαναλάβουμε και να αναμασίζουμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά για να διδαχτούμε κάτι. Το πρώτο λοιπόν μάθημα για μένα ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξή. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια πολιτική κοινών υποσχέσεων και να μείνουν στο κατόφλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης αυτέ οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρή. Αλλά όλοι γνωρίζουμε επίση ότι είναι και δίκαιη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ελέγχθησε σε ό,τι αφορά τις, τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά δεν ήταν δίκαιοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν το 2020 μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Αυτό το δήλωσε στο Ζάγκρεπ η Ούρσλα Φοντερ Λάιεν. Αν θέλουμε να έχουμε μια σωστή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές θεωρώ ότι πολλές είναι οι ευκαιρίε που έχουμε για το 2020, αλλά έχουμε πραγματικά μακρύ δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει να συνεχίσετε τις μεταρρυθμίσεις και να τις πετύχετε με φιλοδοξό τρόπο, να προσανατολιστείτε στις ε, κοινωνίες μας και ω ε, τασμικά όργανα θα πρέπει να ε, εκπληρώσουμε τις υποσχέσει μας. Όταν κάτι λέμε, να το τηρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κούτσοκ και χαίρομαι που βλέπω εδώ τον κύριο Παύλο Ραγγέλ μόνιμο εισηγητή για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τρία λεπτά έχετε ο καθένα σα. Thank you very much. First, I would like to apologize. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας, διότι με ε, απήγαγε ο πρόεδρος της ομάδας μου και ήμουν μαζί του την τελευταία ώρα και έτσι δεν μπόρεσα να είμαι εδώ στην ώρα μου. Θα προετοιμάζαμε μάλιστα κάποιες πτυχές της συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης, όπου ελπίζουμε πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε όλες τις βαλκανικές χώρες. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα ήταν μια πολύ καλή προοπτική για να ξεκινήσουμε γιατί αν σκεφτόμαστε το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορούμε να σκεφτούμε το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τα Βαλκάνια. And so uh, this would be my statement. Χωρίς την... τα Βαλκάνια η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Αυτή, αυτό θα μπορούσε να είναι το, το κυρίως νόημα. Ε, πιστεύω ότι για τη Βοσνία Ζεγοβίνη έχω φέρουμε τεράστια ευθύνη ως Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να βοηθήσουμε να συνεργαστεί ε, να συνεργαστούμε με ισότιμο τρόπο, χωρίς πατερναλισμό, όλους τους ε, διαφερόμενους φορείς, όλους ε, τους θεσμούς, ώστε να αναπτύξουν τις προσπάθειές τους και να μπορέσουν να τηρήσουν κριτήρια και στάνταρ που θα λειτουργήσουν ως ένα πρώτο βήμα για την Βοσνία Ζεγοβίνη ως υποψήφια χώρα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αγωνιστεί γι' αυτό και βεβαίως χρειαζόμαστε τους Βόσνιους φίλους μας για να μας βοηθήσουν γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα όπου πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο και πιστεύω πως αυτό είναι εφικτό. Πιστεύω λοιπόν πως οι Βόσνοι πολίτες από όλες τις κοινότητες αξίζουν την προσπάθεια από πλευράς των πολιτικών, τόσο των Ευρωπαίων όσο και των Βοσνίων. Αξίζουν την προσπάθεια όλων μας για να ε, τους δώσουμε αυτή την προοπτική της σταθερότητας για το μέλλον. Είμαι λοιπόν ε, αισιόδοξος και θετικός ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το επεισόδιο της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελβανίας. Θα είναι ένα επεισόδιο μόνο που ε, ε, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα μπορέσουμε να πούμε πώς πρέπει να δούμε τα Βαλκάνια με θετικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Τάνια Φαγιόν που είναι ε, συμπροέδρος στην Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Σερβία. Ευχαριστώ τον Νίνο. Καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσω σλοβενικά σήμερα διότι μπορώ. Έχουμε διερμηνεί σήμερα εδώ. Εγώ υπηρετώ ως Ευρωβουλευτής εδώ και 11 χρόνια και είναι πρώτη φορά που βλέπω αυτή τη σπουδαία σύναξη όλων των προέδρων του Κοινοβουλίου ολόκληρης της περιοχής ε, ε, των Δυτικών Βαλκανίων είναι ε, μέγα επίτευγμα του Προέδρου Σασόλη, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Το 2020 θα είναι σημαντική χρονιά γιατί μπορούμε να μετατρέψουμε και πάλι τη διεύρυνση σε ε, επιτυχία. Μπορούμε λοιπόν να δουλέψουμε πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και οι πολιτικοί στα Δυτικά Βαλκάνια να μπορέσουν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Ελπίζουμε λοιπόν πως έτσι θα είναι σπουδαία η χρονιά ε, αν όλα δηλαδή αυτά προχωρήσουν προς τη σωστή ε, κατεύθυνση. Το ψήφισμα για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ήταν μεγάλο σφάλμα και για το κοσυφοπαίδιο γιατί το Κωσυφοπαίδιο ήταν ε, η πρώτη χώρα που εφάρμοσε ο, τις μεταρρυθμίσεις και ακόμα περιμένει. Μεγάλα λάθη αυτά ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε πολύ από την αξιοπιστία της λόγω αυτών. Ελπίζουμε πως ε, θα μπορέσουν όλα αυτά να διορθωθούν και πραγματικά ελπίζω ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας ότι όλοι πιστεύουν πως οι προϋποθέσεις για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στηρούνται. Δεν θέλω να δω διαμαρτυρία στους δρόμους, δεν θέλω να δω ε, την απουσία της αντιπολίτευσης από τις εκλογές, δεν θέλω να δω ε, δυσλειτουργικά κοινοβούλια με την αντιπολίτευση στους δρόμους δηλαδή. Ελπίζω ότι Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει θετικά μηνύματα στα Δυτικά Βαλκάνια ώστε να συνεχίσουμε να ε, προχωρούμε. Κάποιος είπε σήμερα ότι όταν η Κροατία ε, ε, δούλεψε σκληρά ανταμείφθηκε. Αυτό είναι αλήθεια αλλά στους προηγούμενους μήνες είδαμε ότι δεν πάνε όλα πάντα ε, κατευχήν. Ε, χρειάζεται μια νέα πνοή, μια νέα δυναμική και ελπίζω ότι μέσα από τη συνεργασία μας και μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάπως περισσότερη υπομονή, πράγμα που θα οδηγήσει και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και έτσι θα μπορέσει να να προχωρήσει και η ε, διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επανέλθει η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην, ε, περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και εμείς πρέπει να είμαστε πιο αξιόπιστος εταίρος γιατί έτσι θα έχουν εμπιστοσύνη και οι πολίτες. Ε, Ούτω ή άλλω, όλοι μας βρισκόμαστε στην Ευρώπη, πρέπει να συνεργαστούμε θετικά και ειλικρινά. Υπάρχουν διάφορα ε, στραβά, αλλά δεν θα πρέπει να παίρνουμε τις επικρίσεις αρνητικά, αλλά ως επικοδομητική κριτική. Ευχαριστώ. Μιλήσατε όλοι οι πρόεδροι και Τώρα το βασικό μας πρόβλημα είναι ο, προϋπολο... είναι χρόνος, γιατί τα επόμενα δέκα λεπτά οι διερμηνείς μας ε, θα ε, τελειώσουν. Γι' αυτό ε, αποφάσισα να δώσουμε λίγο χρόνο σε άλλα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά παρακαλώ να περιοριστείτε στα δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σας. Η κυρία Ζόνκο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά, Πρόεδρε, για να γίνω πιο κατανοητή. Καλώς ήρθατε στη συνάντηση. Ευχαριστούμε που διοργανώσατε τη χρησιμότατη αυτή η συνάντηση σήμερα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας που είπε ότι αυτό το ψήφισμα για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία ήταν φως για σας μια κρίσιμη στιγμή, ακτίδα φωτός μετράνε αυτά τα ψηφίσματα. Αυτό πιστεύουμε. Διαπραγματεύτηκα το ψήφισμα για τη Βόρεια Μακεδονία, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήμουν επικεφαλή των διαπραγματεύσεων για το ψήφισμα για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Είχαμε υποστήριξη από πάνω από 500 ε, συναδέλφους στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε επί προεδρία ε, να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις Και θέλω πράγματι αυτό να συμβεί. Με απασχολεί. Είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση που επικρατεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα αναφέρομαι στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η φωνή του Ευρωκοινοβουλίου ακούγεται εκεί. Αλλά οι αποφάσει δεν εφαρμόζονται. Στην περίπτωση τη βόρεια Μακεδονία, κάτι κάνετε. Στην περίπτωση τη Σερβία και του Μαυροβουνίου και του Κωσυφοπεδίου ακούτε. Αλλά τι συμβαίνει με τη, με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Τέσσερα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου έχουμε σχετικά με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Είχαμε διαπραγματευτεί, διαπραγματεύσει τον Brexit. Αύριο ψηφίσουμε για τον Brexit. Είχαμε την Παρασκευή της μεγάλη Παρασκευής, την ελευτική διαδικασία και φροντίζουμε για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στη Βόρεια Ιρλανδία. Τι γίνεται με το 1 εκατομμύριο Κροάτες πολίτες που ζουν στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Κύριε Σβίτζιτς και κύριε Τζόβιτ, μπορείτε να μας πείτε πότε θα εφαρμόσετε τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βοσνία Ζεγοβίνη, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκρός έχει το λόγο. Τιμή. Δεν ζήτησα το λόγο. Θα μιλήσω κι εγώ σλοβενικά. Έχουμε διερμηνία. Έχουμε, έχουμε, έχουμε. Θα ήθελα να πω ότι προέρχομαι από μια χώρα που υποστηρίζει ένθερμα την ενταξιακή διαδικασία για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πω κάτι επιπλέον, ότι ενδιαφέρομαι και εγώ, διότι προεδρεύω της διακοινοβουλευτικής ε, ομάδας για τη Βοσνία-Ζεγοβίνη θα ήθελα να εφαρμόζετε αυτά που λένε τα ψηφίσματά μας, αλλά αναμένω από εσά να εφαρμόζετε και δικαστικές αποφάσεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όχι μόνο των εθνικών δικαστηρίων, αλλά και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα Βαλκάνια είναι σημαντική περιοχή και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πρόκληση. Συχνά δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε το εξή πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σαφή πολιτική που θεστιάζεται επί συγκεκριμένων χωρών. Αυτές οι χώρες είναι σε διαφορετικά στάδια ετοιμότητας και θα πρέπει να είμαστε και εμείς προσαρμοσμένοι στις διάφορες καταστάσεις, να βοηθάμε τις χώρες ε, να εφαρμόζουν σωστά τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται. Κάποια μέτρα λαμβάνονται ε, λόγω ημών, όπως η μετανάστευση. Ε, η πολιτική για μετανάστευση οδηγεί σε διαχείριση της μετανάστευσης και αυτό είναι υποφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, όχι μόνο για τη γωνία, αλλά τελικά και εσείς ωφελείστε. Εκπροσωπείτε πολλές χώρες και κάποια στιγμή όλοι θέλουμε να σας δούμε να είσαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να αναπτύξουμε κατάλληλους μηχανισμούς που θα σας επιτρέψουν να συμμορφωθείτε, να εκπληρώσετε αυτό το στατικικό ε, ε, στόχο. Βάλκα Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ και σας ε, καλωσορίζω στην διάσκεψη αυτή. Για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι πλήρη όσο κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα λοιπόν θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ε, διεύρυνση και με τι χώρες των Βαλκανίων και με τα Μολδαβία κτλ. Ξεκινήσε λοιπόν η επανάσταση στη ώρα και είχαμε ε, επαφές με το προξενείο της ε, Ιουκοσλαβίας ως Ρουμάνος λοιπόν πρέπει να σας πω ότι σας ενθαρρύνουμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές που χρειάζονται. Όλοι θα πρέπει να σέβονται τους ε, κανόνες και ελπίζω και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολιτικοί να θεωρήσουν ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα ευωδώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φραντμποκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, Πρόεδρους των Κοινοβουλίων. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μεγαλύτερος φίλος είμαστε των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, υποστηρίξαμε και την αρνητική απόφαση του Οκτωβρίου. Είναι ένα σαφές μήνυμα αυτό. Ένα μήνυμα συνεργασία προς την ε, περιοχή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αναμένει καλή συνεργασία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις από κοινού προκειμένου να δώσουμε απαντήσεις σε κοινά ζητήματα. Πώς θα εξασφαλίσουμε σωστή διάβρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε τις ε, ευρωπαϊκές αξίες, να τις προωθήσουμε επίσης στις χώρες σας. Θεωρώ λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει κάποιο χρόνο. Η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί. Καταρχά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει πιο πολλέ προσπάθειε για την παροχή υποστήριξη προ τι χώρε σα προκειμένου να υλοποιήσουν τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει, ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών, τη οικονομία, τη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν πρακτικές λύσεις. Βάσει λοιπόν όλων αυτών θεωρώ ότι οι πολίτες σας θα αντιληφθούν με πολύ πιο εντόνο τρόπο την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Και πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή μεταρρύθμισης θα δώσει την ευκαιρία στις χώρες σας να έχουν πρόσβαση και σε άλλα εργαλεία πέρα από τα πρωτεξιακά εργαλεία. Και βάσει αυτών θα μπορέσετε να πετύχετε με πολύ πιο εύκολο τρόπο τελικά τους στόχους σας για να εκπληρώσετε και τις ε, προϋποθέσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Και αυτό για να φροντίσετε και το 80% των ε, νέων που θέλουν να φύγουν από τη χώρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε και τον κύριο Χερμαν Τάτς. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μετάφραση. Μάλιστα. Εφόσον υπάρχει θα μιλήσω ισπανικά. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα και εγώ να πω ότι πρέπει να δώσουμε μια πνοή. Το χτύπημα του Οκτωβρίου ήταν πολύ βαρύ και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διαχειριστούμε αυτή, την, αυτή την αναποδιά που έχει μεγάλο αντίκτυπο στην περιοχή. Εγώ που γνώρισα τα Βαλκάνια σε πολύ χειρότερους καιρούς, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές του 90, πραγματικά χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ και που σας βλέπω όλους εδώ με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα, το ίδιο project. Όλοι γνωρίζουμε εδώ ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα στα Βαλκάνια, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν θανατηφόρο για την Ευρώπη γιατί το ότι μπαίνει εκεί και το ότι βγαίνει από εκεί μας επηρεάζει όλους. Κανείς δεν μπορεί να κοιτά από την άλλη πλευρά και ο χρόνος περνά. Ο χρόνος δεν είναι καλός σύμβουλος, υπάρχουν άλλα συμφέροντα τα οποία φροντίζουν να μην κλείσει αυτή η μαύρη τρύπα. Πρέπει λοιπόν τώρα στην εκλογική αυτή περίοδο που βρίσκονται αρκετές χώρες να δώσουμε κίνητρα για ένα καθαρό δημοκρατικό project το οποίο θα δώσει πνοή στην πρόοδο, θα δώσει πνοή στις μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση. Είναι ένα κίνητρο το οποίο θα πρέπει να έρθει μέσα από τη βοήθεια και τη στήριξη που θα δώσουμε για να, και ενθουσιασμό και πάλι πνοή νέα για αυτό το κεφάλαιο που έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι και πρέπει να το κλείσουμε με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πραγματικά θα ήθελα να επιταχυνθεί φέτος όλη αυτή τη διαδικασία, όπως έλεγε και η κυρία ε, Φαχών που το είπε ότι ναι, είναι απαραίτητος ο ενθουσιασμός. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδροι των κοινοβουλίων εξ ονόματος του Προέδρου της ΑΦΕ του κ. Μακάλιστερ που δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρόν εδώ. Νομίζω ότι είχαμε και ολοκληρώσαμε μια σημαντική συνεδρίαση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργή σας συμμετοχή και για τις εισηγήσεις σας. Πιστεύω πως όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο που θέλουμε να ευοδοθεί και πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να σπρώξουμε την διεύρυνση. Μια σύντομη παρατήρηση στο τέλος. Πριν, ε, σε τρεις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μικρύνει κατά ένα κράτος μέλος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Όμως, όπως και αν είναι το ο Brexit και θα είναι περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία, νομίζω πως είναι ευκολότερο να φύγει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σήμερα ημέρα. Όμως η πολιτική διεύρυνση πρέπει να ξαναμπεί σε σωστή πορεία. Νομίζω πως με αυτή μας τη συζήτηση θα συμβάλλουμε σε αυτό. Ήθελα να σας ξαναδώ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πριν να κλείσω τη συνεδρίαση θα ήθελα επίσης να πω πως δεν έχουμε χρόνο να ε, σπαταλήσουμε πριν από τη διάσκεψη κορυφής του Ζάγκρεμπ πρέπει να μπορέσουμε να εκφράσουμε σαφή και θετική δέσμευση ώστε να αποκαταστήσουμε την ευρωπαϊκή ενότητα σε σχέση με τη διεύρυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σταθερό και ευημερές μέλλον μόνο αν ενισχύουμε αλλήλους και αν βασίζουμε τις σχέσεις μας στην δημοκρατική ε, στο δημοκρατικό έλεγχο και το κράτος δικαίου. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ αγαπητοί πρόεδροι για τη συμμετοχή σας. Σε παρακαλώ επιστρέψτε στις χώρες σας με την ισχυρή αίσθηση στήριξης που προέρχεται όχι από ένα, δύο, τρει ε, μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, την ηγεσία του Ευρωκοινοβουλίου